Bene. Oui. Euh, το πρώτο θέμα είναι το 10. Ε, Εσάς περιμέναμε κύριε Κράμερ και σας δίνουμε και το λόγο. Μέσω συνεργασίας για την πυρηνική ασφάλεια. Έχετε το λόγο κύριε σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που και περιμένατε. Δεν προβλεπόταν να είμαι εγώ το δικό μου με το πρώτο μου σημείο στην ημερησία διάταξη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πυρηνική ασφάλεια και συνεργασία σε σχέση με αυτήν. Πολύ σημαντική με τρίτε χώρε, μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών. Θα προσπαθήσω σε κάποια λεπτά να παρουσιάσω τι έχω συντάξει στην έκθεσή μου, ποια είναι η αφετηρία για αυτά τα θέματα. Πολλές χώρες ασχολούνται με ε, πολιτική εκμετάλλευση της ατομικής ενέργειας, αστική εκμετάλλευση. Για κάποιους στην Ευρώπη αυτό δεν ταιριάζει ίσως ε, σε σχέση με τις ευκαιρίες, ε, σε σχέση με την βιομηχανία μας και τους ερευνητές μας. Για εκείνους όμως που ασχολούνται με προδιαγραφές ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αστική μη στρατιωτική εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας, σκόπιμο είναι να μιλήσουμε για συμφωνίες και συμφωνίες που πρόκειται να συναυθούν. Θα έλεγα καλό θα ήταν για μας την πρόταση της Επιτροπής στο θέμα αυτό να την υποστηρίξουμε σε μεγάλο βαθμό. Ουσιαστικά δύο μόνο ουσιοδέστερα σημεία θα έχω προσθέσει ή κάπως ενίσχυσα περισσότερο. Νομίζω με τα όσα συνέβησαν στη Φουκουσίμα στην Ιαπωνία για άλλη μια φορά καταδείχθηκε πόσο σημαντικό είναι όσοι εκμεταλλεύονται ως πάροχοι ή δημιουργοί πυρηνικών αντιδραστήρων και που λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον να ε, υπόκεινται σε αρχές αδειοδότησης και αρχές ε, εκμετάλλευσης. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς γραμμές και να μην συγχέονται τα πράγματα ώστε πρώτον να μπορούμε να αποφεύγουμε ανθρώπινα σφάλματα και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Επίσης υπογράμμισα ότι δεν θα έπρεπε να συνεισφέρουμε η δημιουργία πυρηνικών αντιδραστήρων να συγχρηματοδοτείται ή να επιδοθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο ως αρρωγή, παρέχοντας συνδρομή, μπορούμε να δράσουμε όταν πρόκειται για την ασφάλεια, την συνεισφορά μας στην ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων. Δύο λόγια μόνο για τα διαδικαστικά θέματα. Εδώ έχουμε διαδικασία διαβούλευσης ως κοινοβούλιο. Αυτό τι σημαίνει. Προτού ληφθεί μια επίσημη απόφαση στο επίπεδο του Συμβουλίου ή αλλού, το Ευρωκοινοβούλιο καλείται να διαβουλευτεί επ' αυτού. Και διαπίστωσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επίσης και το Συμβούλιο με την Ευρατόμ, έχουν διαπραγματευτεί ένα κομμένο και ραμμένο τελικό κείμενο. Η δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθίσταται ανεδαφική πλέον και ξεπερασμένη και δεν θέλω να αγνοήσω την ευκαιρία και πρέπει να δραθώ τη ευκαιρία ότι δεν πρέπει να είναι νόημα αυτού του εγχειρήματο να γίνεται κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να αναμείνουν πρώτα το Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί και μετά να αποφασίσουν. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Τονίζω, πρόκειται για τη συνεργασία με τρίτε χώρε και όχι για το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας στην ίδια την Ευρώπη. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Εδώ πρόκειται για το πώς μπορούμε εμείς να συνεισφέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για την πυρηνική ασφάλεια εκτός Ευρώπης. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για την έκθεση αυτή. Ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζόρνταν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποστηρίξω από πλευράς μου τον συνάδελφο, τον κύριο Κράμερ, που ανέφερε ότι έχει τεράστια σημασία για την πυρηνική ασφάλεια να έχουμε ένα ισχυρό ανεξάρτητο φορέα για την αξιολόγηση και τους ελέγχους. Πολλές βελτιώσεις προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζονται. Υποστηρίζω αυτή την κατεύθυνση φυσικά. Όμως αναμένουν, πρέπει να αναμένουμε ότι θα είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε διατυπώνοντας κάποιες νέες τροπολογίες για να προχωρήσουμε Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να εμπλακεί σε αυτό το έγγραφο, να εμπλακούν θέματα τα οποία δημιουργούν κάποιες αμφιβολίες ίσως όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλείσιμο πυρηνικών αντιδραστήρων. Από την άλλη πλευρά δεν βλέπω να υπάρχει ανάγκη να περιορίσουμε αυτό το μέσο μόνο αποκλειστικά σε εκείνες τις χώρες που έχουν τέτοια προγράμματα και που ήδη κλείνουν πυρηνικούς αντιδραστήρες. Διότι θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να μεριμνήσουμε για το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και για τον καλύτερο συντονισμό που πρέπει να διασφαλίζεται μεταξύ των χωρών εκείνων που έχουν πυρηνικού αντιδραστήρε σε λειτουργία. Εκείνο που βλέπω να λείπει, να απουσιάζει περισσότερο σε αυτήν την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να καλύψουμε το κενό, είναι ένα μεγαλύτερο και ισχυρότερο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου, που θα έπρεπε διαρκώ να ενημερώνεται και σε τακτά διαστήματα να επικαιροποιείται η ενημέρωσή του στα διάφορα θέματα και θα έπρεπε να έχουμε ένα σαφή ορισμό πώς ε, χώρες ε, υψηλού εισοδήματος ε, έχουν ξεχωριστές επιδόσεις. Πρόσθετα για ένα ισχυρό και ανεξάρτητο φορέα ελεγκτικό για τους ελέγχους και την εποπτεία χρειαζόμαστε καλά καταρτισμένο προσωπικό με αντίστοιχες δεξιότητες και ικανότητες που θα έχει επαρκώς καταρτιστεί για το πρόγραμμα μέσα στο πλαίσιο της Ευρατόμ για τα πυρηνικά ζητήματα. Αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο, ως εργαλείο για να προαγάγουμε ένα υψηλότερο επίπεδο αναβαθμισμένης ασφάλειας σε όλα τα κράτη-μέλη, ως υπόδειγμα για, αυτή την, τα, για αυτές τις νέες δοκιμασίες. Κουάδρας. Κύριος Βίνταρ παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Πράγματι, η συνεργασία της Ένωσης με τρίτες χώρες για να βελτιώσουμε τη πυρηνική ενέργεια ήταν ένα βασικό μέλημα της πολιτικής μας σε αυτό το τομέα. Σήμερα το θέμα μας απασχολεί τη στιγμή που στην Ευρώπη υπάρχουν ε, κράτη-μέλη που άλλαξαν ε, τον προσανατολισμό τους σε σχέση με τις πυρηνικές ε, δοκιμές και δεν είναι λίγες οι χώρες εκείνες που ασχολούνται με την κατασκευή πυρηνικών μονάδων Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Μπαγκλαντές και μέσα στα πλαίσια αυτού του κύματος ε, πυρηνικών δοκιμών ανά τον κόσμο, θα πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε οι χώρες αυτές να οικοδομήσουν τις πυρηνικές μονάδες σύμφωνα με τις ε, προδιαγραφές που ισχύουν και για την ε, Ευρώπη. Γι' αυτό δημιουργήθηκε και ένα μέσον για να συσφίξουμε τις σχέσεις μας, όχι μόνο με τις γείτονες χώρες, αλλά και με άλλες χώρες ανά τον κόσμο που θέλουν να παράγουν πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Ο συνάδελφος Κράμερ έχει βελτιώσει το κείμενο και ελπίζουμε ότι στην οδηγία θα συμπεριληφθούν και θα είναι πιο επαρκής η οδηγία. Ενδιαφέρον έχει η βελτίωση της διακυβέρνησης και η ανεξαρτησία των οργανισμών ρύθμισης. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί γιατί στην Ευρώπη έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να είναι ανεξάρτητες αρχές. Γι' αυτό το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και στις τρίτες χώρες. Επίσης, όπως είπε και ο συνάδελφος Κράμερ, θα πρέπει να επιμείνουμε στη διεθνή συνεργασία ως στοιχείο για τη μη διάδοση των πυρηνικών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρότερο πλαίσιο. Ξέρουμε τι συμβαίνει στο Ιράν με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και ο κύριος Κράμερ ε, είναι πολύ εύστοχος σε αυτή τη μνήμα. Όπως αναφέρει και η τροπολογία 6 του εισηγητή, μας ενδιαφέρει η συμμετοχή Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων σε, από τις τρίτες χώρες. Υπάρχουν χώρες που έχουν εγκαταλείψει το πυρηνικό τους πρόγραμμα και άλλες που θα πρέπει να αναθεωρήσουν τη θέση τους μεσοπρόθεσμα. Υπάρχει όμως μεγάλος κίνδυνος να χάσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας μέσα στα πλαίσια της εμπειρογνωμοσύνης στην Ευρώπη και γι' αυτό χρειαζόμαστε νέους εμπειρογνώμονες που να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την τεχνογνωσία για μελλοντική, για μελλοντική χρήση. Ζαντώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τον συνάδελφο Βιντάλ Κουάδρας με μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντα και μίλησε για πυρηνικού σταθμού στον Μπαγκλαντές. Περίεργο. Εγώ έζησα στον Μπαγκλαντές, εργάστηκα για την ε, αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί προσπαθούσαμε φράγματα να κάνουμε στο Μπαγκλαντές. Είχαμε τεράστια ε, διεθνή συνεργασία, δαπανίσαμε 200 εκατομμύρια δολάρια σε μελέτες ε, και εμπειρογνώμονες για να φτιάξουμε φράγματα, υδατοφράκτες, προκειμένου να μην έχουμε πλημμύρες και στη τελική ανάλυση ούτε ένα φράγμα δεν καταφέραμε να κατασκευάσουμε. Γιατί οι κοίτε των ποταμών είναι τόσο ευμετάβλητες και το έδαφος τόσο ε, αμαλακό που δεν μπορούμε ούτε καν ε, την κήτη να διοχετεύσουμε. Και το, μιλούμε τώρα για δημιουργία πυρηνικών σταθμών για μια χώρα που τα δύο τρίτα της ε, κάθε χρόνο βρίσκονται κάτω από το νερό με τεράστιες πλημμύρες. Είναι λάθος να μιλάμε για προοπτική ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας παντού. Λάθος, παρόλο που είμαστε υπέρ της πυρηνικής ενέργειας. Η ευρωπαϊκή εμπειρία τώρα. Φυσικά έγιναν αυτά τα τεστ αντοχής των πυρηνικών σταθμών και ξέρετε ότι η πράσινη ήταν πολύ επικριτική για τις δοκιμές αυτές αντοχής, γιατί δεν έλεξαν υπόψη πολύ κίνδυνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο πυρκαγιάς, ανθρώπινου λάθους, η δολιοφθοράς, κακόβουλης επίθεσης. Ε, αυτό συνέβη και με τους ε, Ιάπωνες. Είδαμε ότι ούτε εκεί υπήρξε ε, επιτυχία σε ό,τι αφορά τη συνεργασία για να μειωθεί ε, ο πυρηνικός κίνδυνος. Και δύο τελευταία σχόλια. Ναι, θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο ότι αφορά την ανεξαρτησία των αρχών πυρηνική ασφάλεια. Είναι επιτακτική ανάγκη. Δεν γνωρίζω το καταστατικό όλων των αντίστοιχων οργανισμών πυρηνική ασφάλεια, αλλά στη Γαλλία τουλάχιστον τα μέλη ορίζονται από τι πολιτικέ αρχέ. Και όταν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο κλάδος των πυρηνικών, η πυρηνική βιομηχανία, είτε στρατιωτική είτε μη στρατιωτική, η πολιτική παρουσία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η άλλη της κυβέρνησης και ο διορισμός, ο πολιτικός διορισμός των μελών του οργανισμού δεν εξασφαλίζει ανεξαρτησία αυτής της ρυθμιστικής αρχής. Σε ό,τι αφορά την κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων σε διάφορες χώρες που μπορεί να οδηγήσει σε διάδοση των πυρηνικών. Όντω είναι πολύ καλή τεκμηρία που μα δίνει ο ΙΕ για τα θέματα αυτά για τον κίνδυνο, γιατί δεν υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ της στρατιωτικής και μη στρατιωτικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Στις Ηνωμένε Πολιτείε επικρατεί ένα σύστημα που λειτουργεί σχετικά εύρυθμα. Όλες οι ευαίσθητες τεχνολογίες και όλες οι πωλήσει ευαίσθητων τεχνολογιών θα πρέπει να περνούν από το Κογκρέσο. Σε ελάχιστες χώρες υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να φανταστούμε κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι στα πλαίσια κατά ανάγκη αυτής της οδηγίας, να εκφέρουμε τη γνώμη μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξαγωγή ευαίσθητων τεχνολογιών και άρα και της πυρηνικής τεχνολογίας προς διάφορες χώρες. Γιατί όταν η Γαλλία ήθελε να πουλήσει το καντάφι στη Λιβύη πυρηνικό εργοστάσιο ένα χρόνο μετά την απόσυρση της Λιβύης από το κατάλογο των χωρών με τρομοκράτες. Μη μου λέτε ότι σκοπός ήταν να δημιουργηθεί πυρηνικό εργοστάσιο για μη στρατιωτικό σκοπό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή που θα ήθελε να σχολιάσει. Όχι, ο κύριος Κράμερ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους <clears throat> για την ευρύτερη υποστήριξη της έκθεσής μου. Φυσικά τροπολογίες ε, πρέπει να κατατεθούν όπου χρειάζεται. Το ότι δεν τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θλιβερό σε σχέση με αυτά που είπα. Ποιο νόημα έχει μια διαδικασία διαβούλευσης όταν συντάσσονται κείμενα που de facto δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη στην πρακτική εφαρμογή και όταν πρόκειται για τη σύναψη ε, συμφωνίας με την Ευρατόμ. Νομίζω ότι τα σημαντικότερα σημεία επί των οποίων συμφωνούμε είναι όλα συνενετικά και το θέμα της διακυβέρνησης και διαχείρισης ε, δεν νομίζω τώρα ότι είναι σκόπιμο εδώ ξεχωριστές χώρες να αναφέρονται ως παραδείγματα. Αυτή η σύμβαση δεν είναι για να μπορεί να υποστηριχθεί η δημιουργία ποινικών αντιδραστήρων στο Μπαγκλαντές. Είναι πολύ τραβηγμένο αυτό το παράδειγμα και πολύ δυσνόητο. Τώρα η συνεργασία στο θέμα αυτό μόνο τότε μπορεί να επιτευχθεί όταν γνωρίζουμε ότι άλλα κράτη είναι ανεξάρτητα στις αποφάσεις που λαμβάνουν για την εκμετάλλευση πυρηνικής ενέργειας και την δημιουργία πυρηνικών αντιδραστήρων. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τέτοιου είδους συνεργασία σε κανένα κράτος. Έχει αρκετά να προσφέρει η Ευρώπη και γι' αυτό το μέσο αυτό το οποίο έχουμε επιτραπέζει σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να βελτιωθεί, να είναι ένα με νόημα, σκόπιμο μέσο για να τύχει υποστήριξη. Έτσι ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λίγη στις 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ, το COP18 δηλαδή. Κυρία Ουλσκοκ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω σου ειδικά. Πολύ σας ευχαριστώ. Πρόκειται για το, την αντιπροσωπεία του ΕΛΚΑ και τη συνεισφορά σε, σχέση με την ε, Σύνοδο για τις ε, κλιματικές αλλαγές ε, αρχές Δεκεμβρίου. Είχαμε εξαιρετικέ συζητήσεις με όλες τις πολιτικές ομάδες και προφανώς γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά το e-trade υπό δική μας αρμοδιότητα. Εμείς ε, έχουμε την αρμοδιότητα. Παραμένουμε λοιπόν σε σχέση με τις δικές μας αρμοδιότητες. Η επόμενη συνεδρία θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου Μέχρι σήμερα έχουμε ένα κείμενο, μπορώ να πω, ένα κείμενο το οποίο βασίζεται στις προηγούμενες συμφωνίες σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Σε αυτά βασιστήκαμε και κάναμε και κάποιες προσθήκες. Κάνουμε λόγο και για την Σύνοδο Κορυφής του Ρίο Ντεζανέιρο. Αυτά όσον αφορά το κείμενο. Κάνουμε επίσης λόγο για την Λέσχη των 20, G20, και που στο Μεξικό, στο Λοσκάμπος, παλήθευσαν, επιβεβαίωσαν προηγούμενες αποφάσεις να πάψουν να υπάρχουν επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις όσον αφορά την εξόριξη ορυκτών καυσίμων. Μπορώ να σας πω ότι το κείμενο κάνει λόγο για εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και για ορυκτά καύσιμα. Ανησυχούμε για αυτά, διότι το 2011 οι εκπομπές ρήπων ε, εις βάρος της ατμόσφαιρας ε, αντί να έχουν μειωθεί έχουν αυξηθεί και αυτό είναι πολύ αρνητικό. Επίσης ε, τονίζουμε ότι πολλές μη ευρωπαϊκές χώρες επενδύουν τεράστια κονδύλια στην ενεργειακή μεταβολή και επενδύουν σε αυτές τις κατευθύνσεις. Ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό για μας, για το δικό μας μέλλον και την ανταγωνιστικότητά μας στο μέλλον. Επίση, κάνουμε λόγο για την χρηματοοικονομική κρίση. Λέμε δεν πρέπει να υπονομεύει στο κατά την δική μα διαπραγματευτική θέση. Και όσον αφορά το ενεργειακό δυναμικό. Εκφράζουμε τη θλίψη μας διότι δεν χρησιμοποιούμε αυτό το ενεργειακό δυναμικό ούτε διεθνώς ούτε από πλευράς ΕΕ ξεχωριστά. Κάνουμε λόγο για τις αγορές και για νόμους για τη διαμόρφωση των τιμών και λέμε ότι όταν πρόκειται για την αλλαγή ενεργειακής εκμετάλλευσης πολλοί δεν ευθυγραμμίζονται όπως θα έπρεπε. Υπάρχουν διάφορες περιπλοκές. Όλοι, όλες οι πολιτικές ομάδες εμπλέκονται και θα ήθελα να διασφαλίσουν ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στη Σύνοδο για τις κλιματικές αλλαγές με ένα καλό κείμενο που όλοι μπορούμε να πούμε ότι μας εκπροσωπεί και αντανακλά τις θέσεις μας. Εδώ όπου χρειάζεται φυσικά τίθενται θέματα συμβιβασμών που πρέπει να επιτευχθούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Ζαντό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία θα ήθελα να επενέσω την εισηγητρία για το πολύ αξιόλογο απόνημά της και την ε, προσπάθεια με διαλαξία και επικοδομητικότητα να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις. Δεν περιμέναμε την έκθεση αυτή τόσο γρήγορα. Ήδη γίνεται λόγος για κάποιες ε, για κάποια διαφυγή άνθρακα, carbon leakage, δυνατότητα δηλαδή με την κατάσταση πολλών βιομηχανιών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν φανταζόμασταν ότι αυτές οι μετακαταστάσεις θα λάβουν χώρα τόσο γρήγορα και σε μάλιστα σε τομέα όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ευρώπη είχε ανέκαθεν να αντιμετωπίσει μια πολύ ισχυρή, ένα πολύ ισχυρό ανταγωνισμό και αθέμητο εκ μέρους της Κίνας που μαζικά αύξησε τις παραγωγικές της δυνατότητες. Βέβαια έτσι εξυπηρετούνται οι στόχοι της για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά μιλούμε ουσιαστικά για μια στρατηγική κατάκτηση της διεθνούς αγοράς. Ήταν έντονη η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών με, με τελωνιακούς δασμούς μέχρι 135%. Όταν τα αναφέραμε αυτά τα θέματα με τον, προς τον Επίτροπο και τον πρόεδρο Μπαρόζο έδειξαν ότι ανησυχούν και προβληματίζονται, ε, συναφριώθηκαν, αλλά από ουσιαστική άποψη δεν έχουμε καμία πραγματική στρατηγική για να δούμε αν θέλουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή βιομηχανία και κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργεια που θα είναι καινοτόμο και θα βρίσκεται εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, επαναλαμβάνω, είμαι υπέρ της έκθεσης, αλλά θα ήθελα να κάνω και μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι απαράδεκτο σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να σιωπεί και να ε, παρακολουθεί με σταυρωμένα χέρια ε, φορτία φωτοβολταϊκών που δεν μπορούν να εκφορτωθούν στις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά θα καταφτάσουν στο Ρότερνταμ ε, στο Άμστερνταμ και θα είναι κινέζικες προέλευσης. Έχουμε τη ε, δυνατότητα να αντιδράσουμε για να προστατεύσουμε τη δική μας φωτοβολταϊκή βιομηχανία. Ευχαριστώ. Κυρία Χίμπνερ, σας ευχαριστώ. Ε, πλησιάζει η επόμενη διάσκεψη κορυφής, μια διάσκεψη κορυφής που θα μετατρέψει το κέντρο βάρους από την προστασία του περιβάλλοντος σε θεωρητικό επίπεδο σε μια έμπρακτη προστασία περιβάλλοντος και όχι μόνο με μη δεσμευτικού κανόνες. Είναι σημαντικό για την πολιτική μου ομάδα οι προτινόμενες ε, συμφωνίες και προτάσεις ε, να γίνουν δεκτές σε διεθνές επίπεδο. Γιατί όλα τα μέχρι τώρα βήματα που έγιναν στις διαδοχικές συναντήσεις και διασκέψεις κορυφής δεν είχαν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα γιατί ουσιαστικά υπαναχωρήσαμε και δεν είπαμε τι μπορούμε να συμφωνήσουμε από κοινού και τι έγγραφο ε, μπορούμε να προωθήσουμε ως δεσμευτικό, αλλά για ολόκληρη τη, ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί χωρίς οικουμενική παγκόσμια συμφωνία δεν έχει κανένα νόημα να μιλούμε για τις δικές μας δράσεις και για τις δικές μας προσπάθειες που θα είναι ε, περιορισμένες μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι νευραλγική σημασία σε αυτή η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών να γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και η πίεση που θα ασκήσουμε να είναι για μια συμφωνία οικουμενική, παγκόσμια και όχι μόνο ευρωπαϊκή. Ένα άλλο σημείο σημαντικό, ότι σήμερα μέρα που αντιμετωπίζουμε σοβαρότατη κρίση. Δεν ξέρουμε πώς θα προδιαγραφεί το μέλλον. Αλλά σήμερα δεν μπορούμε να αφήνουμε για το μέλλον τις προσπάθειες μείωσης. Δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε τους στόχους που είχαμε ε, στο παρελθόν, αλλά θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη και την ε, οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε και Μπορεί να συσσωρεύουμε τη μία πρόκληση μετά την άλλη, αλλά αυτές οι προκλήσεις είναι μόνο στα χαρτιά. Έχουμε ήδη κάποιες προτάσεις ε, για επίπεδα μείωσης, αλλά προσοχή να μην αποβούν αυτά τα ποσοστά εις βάρος της ε, κοινοτικής βιομηχανίας, για να μην έχουμε μετεγκατάσταση των βιομηχανιών εκτός των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. μάλλον που αν ε, χάσουμε την παραγωγή και μετα... μετεγκατασταθεί αυτή η βιομηχανία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν πρόκειται να μειωθούν τα επίπεδα των καυσέριων. Θα υπάρξουν εκπομπές καυσέριων, απλώς θα γίνουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την Ρωσία, σίγουρα αναπτύσσεται μια βιομηχανία. Φυσικά όλοι οι άνθρωποι θέλουν να απολαύσουν την ευημερία που δίνει ο πολιτισμός και οι τεχνολογίες. Σίγουρα θα χρειαστούν νέες ε, και περισσότερη ενέργεια. Ίσως όμως, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ίσως υπάρξει άξιο των εκπομπών. Αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε αυτό το επίπεδο των εκπομπών και για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους θα πρέπει να στραφούμε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και νέων λύσεων που θα είναι καινοτόμε και που θα χρησιμοποιούν αποτελεσματικέ τεχνολογίες ε, ορυκτών καυσίμων, θα αναπτύσσουν καλύτερες ε, τεχνολογίες, καλύτερες ενεργειακή απόδοσης, ε, μη συμβατικές μορφές ενέργειας επίσης να αναπτυχθούν, ώστε να έχουμε ένα σωρευτικό αποτέλεσμα να μπορούμε ανα πάσα στιγμή να χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια. Τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει σήμερα και γνωρίζω ότι τέτοιου είδους καινοτομία θα έδινε ευκαιρία και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά και θα έδινε την ευκαιρία στην Ευρώπη για βιώσιμη ανάπτυξη. Άλλο σημαντικό θέμα που θα ήθελα να επισημάνω είναι το πολύ σημαντικό θέμα των εισαγόμενων εκπομπών. Με βάση την έκθεση του Βρετανικού Κοινοβουλίου, σε ό,τι αφορά το outsourcing των εκπομπών, οι εκπομπές από εισαγόμενα προϊόντα αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από τις εκπομπές των δικών μας προϊόντων. Αυτό είναι ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο και δεν είναι γνωστό πολλές φορές. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει από τώρα να το διευθετήσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζόρνταν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε χρόνο προετοιμάζουμε ένα τέτοιο ψήφισμα και πάντα έχουμε μια πρόκληση που αντιμετωπίζει ο εισηγητής. Τι θα πρέπει να προσθεθεί σε αυτό το ψήφισμα για παράδειγμα. Νομίζω είναι σαφές ότι οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη φιλοδοξία για την μείωση εκπομπών ρήπων δεν θα μπορεί να αναμένεται ως αποτελεσματικό στοιχείο Καινοτόμε δράσεις μπορούν να αναμένονται ότι θα προσθεθούν φέτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ακόμα την κρίση και οι δυσκολίες ε, μεγεθύνονται, ενώ η Κίνα καθόλου δεν ε, ανταποκρίνεται. Και ίσως ε, θα πρέπει να διερωτηθούμε ποια είναι τα μετρήσιμα αποτελέσματα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι Κίνα θα έπρεπε να ξεκινήσει να φέρεται με πιο υπεύθυνο τρόπο και ότι θα έπρεπε να υπομειστεί ένα ευρύτερο μέρος των ευθυνών και του βάρους. Αυτό σαφώς θα πρέπει να αναφέρεται στο ψήφισμά μας. Θα έπρεπε ουσιαστικά να απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο φιλόδοξη και να, έχει, να θέσει υψηλότερα τον πύχη σε όλες τις διαπραγματεύσεις και τις σε παγκόσμια κλίμακα προσπάθειες που καταβάλει η σημασία, η σπουδαιότητα δόθηκε μέχρι σήμερα στα στους στόχους που θέσαμε οι ίδιοι ενώπιόν μας στα προγράμματά μας. Όμως οι διεθνείς μας προσπάθειες θα πρέπει να ενταθούν σε αυτό το πλαίσιο, διότι όλες οι κλιματικές αλλαγές είναι παγκόσμιου χαρακτήρα, παγκοσμιοποιημένες και οι λύσεις πρέπει και αυτές να έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα και να είναι και αυτές παγκόσμιες. Σημείωσα σε αυτή την έκθεση και κάτι άλλο, το ότι επαναλαμβάνουμε το ότι θα έπρεπε λέει να είμαστε σε θέση να μειώσουμε τις εκπομπές τρύπων χωρίς να χάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Όμως, εφέτος είναι η χρονιά που θα έπρεπε να αποφύγουμε τέτοιου είδους διατυπώσεις διότι είναι ένα γεγονός το οποίο αναγνωρίζουμε ότι η ΕΠΑ και η Κίνα πολύ περισσότερο προσαρμόστηκαν στους όρους αυτής της κρίσης. Ας μην τα λέμε εμείς με τέτοιου είδους διατυπώσεις στο ψήφισμά μας εφέτος τουλάχιστον. Διότι αυτό θα το πάρουμε για τις διαπραγματεύσεις. Ας μην τους δώσουμε πρόσθετα επιχειρήματα εναντίον μας λοιπόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζόρταν έχει δίκιο. Όλες αυτές οι σωρία ψηφισμάτων μου θυμίζουν τον Τζόνι Λόγκαν. Γιατί κάθε χρόνο ακούμε τα ίδια και τα ίδια Θέλουμε μια διεθνή δεσμευτική συμφωνία όχι μόνο για το κλίμα, αλλά για να υπάρχει και ίση πρόσβαση στην ανταγωνιστικότητα. Κάθε χρόνο όμως είναι ολοένα και πιο δύσκολο να πιστεύουμε να πιστέψουμε σε αυτό το εγχείρημα. Ίσως το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για το κλίμα είναι να σταματήσει όλη η διαδικασία έτσι ώστε να κάνουμε μια οικονομία, μια εξοικονόμηση στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για συμφωνία με την Κίνα και τη ΣΥΠΑ. Γιατί η Κίνα να παραβεί ένα βασικό κανόνα που διέπει τις εξωτερικές της σχέσεις γιατί να δεσμευτεί διεθνώς και με ένα μεγάλο κίνδυνο να μην είναι αξιόπιστη όταν το Αμερικανικό Κογκρέσο έτσι και αλλιώς απορρίψει αυτή τη συμφωνία. Ίσως θα πρέπει να δούμε εναλλακτικές πορείες και να βασιστούμε στην αγορά για να προχωρήσουμε γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόοδο σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών μέσα στα πλαίσια μεμονωμένων κρατών και περιφερειών. Γι' αυτό θα πρέπει να συντονίσουμε αυτές τις προσπάθειες με βάση την αγορά, τις δυνάμεις της αγοράς μπορούμε να ακολουθήσουμε τις καλύτερες περιπτώσεις, τις καλύτερες πρακτικές, να έχουμε τομεακές προσεγγίσεις και να προωθήσουμε τεχνολογία και την καινοτομία. Αυτές τις ε, εταιρικές σχέσεις. Γι' αυτό θα ξεφύγουμε από την ιχνηλάτηση των Ηνωμένων Εθνών και θα υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στα προγράμματα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστούμε το συνάδελφο Ρόντε, η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αυτό που θα ήθελα ε, θα ήταν να κάνω μια επισκόπηση το μέχρι τώρα διαπραγματεύσεων και το τι αναμένεται για τον Μάιο, γιατί στον Τέρμπαν ουσιαστικά σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει με την Κίνα. Και το 2015 θα έχουμε μια παγκόσμια συμφωνία με στόχο τη σημειώσει μέχρι το 2020. Φέτος είναι μια σημαντική χρονιά, μπορεί να είναι μια ακόμη χρονιά, αλλά θα πρέπει να προγραμματίσουμε τη διαπραγματευτική μας τακτική και τη μορφή του νέου καθεστώτος ώστε να εξασφαλίσουμε τη νομική του δεσμευτικότητα για όλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες. Βέβαια, μια τετραετία φαίνεται μακρύ χρονικό διάστημα, αλλά είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε από φέτος με πολύ γερά θεμέλια. Στον Τέρμπαν συμφωνήθηκαν τέσσερα βασικά στοιχεία. Καταρχήν, δεχόμαστε δεύτερη ε, ε, περίοδο δέσμευση από το χρόνο, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα προχωρήσουν σημαντικά προς μια νομικά δεσμευτική συμφωνία και επίσης θα ε, μειώσουμε τη διχοτόμηση μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών σε τη φορά της αναλήψης υποχρεώσεων και επίσης ε, να αυξήσουμε τις δεσμεύσεις μας και πριν το 2020. Είναι εξίσου σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι συμφωνήσαμε για δεύτερη δέσμευση, περίοδο δέσμευση ό,τι αφορά το πρωτόκολλο του Κιώτο και αυτό είναι ένα τμήμα του πακέτου. Υπό τον όρο ότι και οι υπόλοιποι θα υλοποιήσουν καλόπιστα αυτά που συμφωνήσαμε στον Τέρμα και όντω θα σημειώσουμε πρόοδο προς μια νομικά δεσμευτική συμφωνία. Το Μάιο ε, είχαμε όντως κάποια παραχώρηση ορισμένων χωρών που φαίνεται ότι θέλουν να ξανατεθεί επιτάπητο στο πακέτο. Αυτό είναι συνηθισμένο γιατί μπορεί οι υπουργοί να συμφωνούν σε κάτι αλλά οι γραφειοκράτες μετά να παλινδρομούν. Θα πρέπει να αποτρέψουμε αυτή την επαναχώρηση και πραγματικά να εφαρμόσουμε τα συμφωνηθέντα πέρυσι. Από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντικό και αναφέρθηκε και από ορισμένα μέλη της Επιτροπής σας ότι χρειάζεται μία αύξηση των φιλοδοξιών μας. Βέβαια φέτος θα είναι πολύ δύσκολο να αυξηθούν οι φετινές προσφορές, αλλά θέλουμε και συμπληρωματικές πρωτοβουλίες, ήδη ξεκίνησαν για τις, α, τη σπήρωση των δυνάμεων για τις κλιματικές αλλαγές και θα πρέπει να συνεχίσουμε και διμερείς συνεργασίες παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις των ΟΗΕ. Γιατί οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι πολύ συχνά χρονοβόρες και επίμονες. Αλλά δεν υπάρχει ανεναρακτική. Ε, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να στερηθούμε, παρόλο που μπορούμε να διερευνούμε και άλλες οδούς διαπραγματεύσεων και λύσεων. Ευχαριστώ εισηγητής. Η κυρία, η συγκεντρία μάλλον, η κυρία Ούλσκοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες για τις προτάσεις και σχόλια και παρεμβάσεις σας. Τα πράγματα έχουν ως εξή. Δεν θα αναδιατυπώσουμε το ψήφισμα. Δεν θα ανασυντάξουμε από ένα χρόνο στο άλλο το ψήφισμα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε και είναι σημαντικό είναι να διατηρήσουμε τις ε, δικές μας ε, θέσεις και το μήνυμά μας. Το κύριο μήνυμά μας είναι ότι θέλουμε να έχουμε φιλόδοξους στόχους, θέλουμε να υπάρχει μια συμφωνία κοινή, δεσμευτικού χαρακτήρα συμφωνία. Αυτά είναι αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε και για αυτούς τους λόγους πρέπει Διαρκώς να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε. Πρέπει να περνάει το, μήνα, το μήνυμα αυτό στους εταίρους μας κάθε χρόνο εκ νέου. Αυτοί που εργάζονται και συνεργάζονται αυτή την προσέγγιση για το ψήφισμα, όπως γνωρίζω, συμφωνούν από αυτόν. Δεν θέλουμε να εισαγάγουμε δραματικές αλλαγές. Δεν είναι αυτό η ουσία. Αυτό που κάνουμε φυσικά είναι να λαμβάνουμε υπόψη τα τεκτενόμενα γύρω μας από την τελευταία φορά που διατυπώσαμε ένα τέτοιο κείμενο και γι' αυτό κάποια πράγματα συμπληρώνουμε, κάποια άλλα τα ολοκληρώνουμε λαμβάνοντα υπόψη τις πρόσφατες ε, εξελίξεις ώστε να έχουμε ένα κείμενο που όλοι μπορούμε να υποστηρίξουμε. Αυτή είναι η προσέγγιση και έτσι εργαζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι εργαζόμαστε και μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Και όλα όσα γίνονται βέβαια στα Ηνωμένα Έθνη είναι περίπλοκα. Δεν κάνουμε λόγο μόνο για 27 κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει όμως άλλη εναλλακτική λύση από αυτήν. Καμιά φορά μπορεί να ακούγεται σαν μια άλλη επιπλέον χρονιά επανάληψης όλων αυτών και ίσως ε, μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά θα ήθελα να σας πω ε, από τον Durban πρέπει να δούμε ότι έχουν κάποια πράγματα προχωρήσει. Επιστρέφοντας από αυτές τις ε, συνόδους κλιματικών αλλαγών λέμε καμιά φορά δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα, δεν προχωρήσαμε όπως θέλαμε Ίσως επειδή ακριβώς δεν πετύχαμε όλα όσα θέλαμε, όμως τουλάχιστον επιτυγχάνεται κάποια πρόοδος και στην τελευταία σύνοδο στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής ήταν σαφές ότι στο τέλος τέλος είχαμε μια συμφωνία μεταξύ ΙΠΑ και Κίνας που επετεύχθη. Μια συμφωνία που δεν ήταν σύμφωνα με τις απόψεις μας επαρκώς φιλόδοξη και ε, θα έλεγα ικανοποιητική, αλλά παρόλα αυτά ήταν μια συμφωνία και όσον αφορά το βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικό μας βάρος ήταν ε, σημαντικό, είχε αποφασιστικό χαρακτήρα. Όλη η όθηση και η ενεργητικότητα προερχόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δώσαμε τις μεγαλύτερες τέτοιες ε, τοποθετήσεις και πιο έντονες τοποθετήσεις για να προαχθούν αυτά τα θέματα. Ίσως δεν ανταποκρίνονται στις υψηλότερε φιλοδοξίες μας, αλλά παρόλα αυτά ήταν ένα κάποιο αποτέλεσμα και αυτό μετράει. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν, να διασφαλίσουμε και να συνεχίσουμε τις φιλοδοξίες μας, να συνεχίσουμε να στοχεύουμε ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο συνενετικό και ομοθυμίας ώστε να μπορέσουν αυτά τα θέματα να προαχθούν όσον αφορά τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα Ηνωμένα Έθνη. Οι πολιτικές κλιματικές αλλαγές δεν επιτυγχάνεται μια νυχτή. Δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό αλλά παρόλα αυτά έχει σημασία υπαρξιακή για μας, ε, για την επιβίωσή μας και γι' αυτό είναι σαφές ότι πρέπει να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να πετύχουμε σε αυτό με τη συμφωνία μας. Ευχαριστώ χωρίς να ε, ακολουθήσω τους κανόνες, θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Ζαντό ζήτησε το λόγο για δεύτερη φορά. Ε, εκτάκτος σας τον δίνω. Νομίζω ότι η Επιτροπή δεν μας απάντησε πλήρως, γιατί και η Γαλλία θα ήθελε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, αλλά εγώ ασχολούμαι με τη βιομηχανία, όχι το περιβάλλον. Σε σχέση με τις ε, κινέζικες εισαγωγές δεν έλαβα απάντηση από την ε, Κομισιόν, ούτε από την Κομισιόν, ούτε από την εισηγήτρια. Η Κομισιόν έχει κάτι να πει ή θα το αφήσει έτσι. Ό,τι νομίζετε. Ευχαριστώ. Σημειώσαμε το σχόλιο σας, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε με τους συναδέλφους που ασχολούνται και με εμπορική πολιτική. Δεν είναι μόνο θέμα κλίματος, πάντως ε, το σημειώσαμε. Προχωρούμε. Περνάμε στο σημείο που αφορά την ενεργειακή απόδοση και κατάργηση οδηγιών, δύο οδηγιών. Το λόγο έχει ο κύριος Τούρμες. Έχω και ένα διαδικαστικό πριν ξεκινήσουμε την κατουσία συζήτηση. Εγώ ε, είχα καταλάβει, όπως και σκιώδεις ότι η συζήτηση θα ξεκινούσε στις 5. Αυτό είχαμε προγραμματίσει. Οπότε προτιμώ να μην ξεκινήσουμε δεν είναι παρόντες ε, οι Κότ, Χολ και Τόμσον, οι σκιώδεις συγητές. Αλλιώς θα πούνε ότι ήταν άδικο. Μετατοπίσαμε τη συζήτηση νωρίτερα και θα, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος. Έπρεπε να το είχαμε διευκρινίσει. Να μην πούμε τα οι ότι ήταν παρόν μόνο οι και δεν είχαν την ευκαιρία εκείνη να μιλήσουν. Είναι η τελευταία συζήτηση ε, πριν τις ε, διακοπές. Προτιμώ να κάνω μια πεντάλεπτη διακοπή, να τηλεφωνήσουμε τους σκιώδεις ηγητές, αν πρόκειται να έρθουν να τους περιμένουμε, γιατί τέλος θα είναι άδικο. Και το λέω, γιατί το πρώτο που σημείο θα είναι θερμές ευχαριστήσεις προς όλους τους σκιώδεις ηγητές για την ε, τεράστια προσπάθεια που έκαναν να μην δημιουργηθεί η... ένα αρνητικό κλίμα μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και του εισηγητού. Κρίμα Απλώς ήθελα να υπενθυμίσω στον συνάδελφο Τούρνες ότι η ημερήσια διάταξη δεν προβλέπει ωράρια. Ωράρια προβλέπονται μόνο για τη συνάντηση των συντονιστών. Όλα τα άλλα έπονται, δηλαδή έπεται το ένα του άλλου. Δεν ε, θέτουμε ωράρια. Οράρια υπάρχουν μόνο ενδεικτικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχουν, δεν προβλέπονται. Η Πιλάρντε Καστίγιο έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να απογοητεύσω τον αγαπητό συνάδελφο Κλοντ, αλλά Δεν νομίζω ότι τα όνοματα οι βουλευτέ που ανέφερε βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, στο κτίριο, για ευνόητου λόγου. Αλλά α ξεχάσουμε ότι θα έρθουν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι ειδοποίησαν ότι δεν θα έρθουν ούτω ή άλλω. Ο Μάρκο Πίπερ, για παράδειγμα, που είναι σκιώδη ηγητή του ΕΛΚ, ήδη δήλωσε ότι κολλείεται. Γι' αυτό και μου ανέθεσε να εκφέρω εγώ τη γνώμη του εκ μέρου ομάδα, αλλά επιγραμματικά γιατί νομίζω ότι έγινα δεκτά τα περισσότερα σημεία, όχι όλα φυσικά. Κλοντ, αυτή είναι η στιγμή πραγματικότητα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στη συζήτηση. Είναι σημαντικό να μας υπεθυμίσει τα πολύ αξιόλογα επιτεύγματα και με τη δική μου παρέμβαση σας δίνω ήδη το, την κατευθυντήρια γραμμή. Λέω ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό και ότι είχαμε μία μεγάλη ομόνια και συσπηρωμένη θέση, συντεταγμένη που ήταν κέρια σημασία για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα που καταλήξαμε και να επιτύχουμε αυτά που επιτύχαμε. Αλλιώ δεν θα τα καταφέραμε. Είχαμε πολλέ ευκαιρίε να συζητήσουμε το θέμα αυτό και στην Επιτροπή μα αλλά και εντό των πολιτικών ομάδων. Ήδη στην δική μου πολιτική ομάδα συζητήσαμε αυτό το θέμα εκτενέστατα. Φαντάζομαι και οι υπόλοιπε ομάδε το ίδιο έκαναν. Οπότε, δεδομένη τη στιγμή, καλό θα ήταν να συζητήσουμε τώρα το θέμα, ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να γίνει εκτενή συζήτηση. Και τις ευχαριστήσεις, μην ανησυχείτε, θα τις μεταβιβάσουμε στους ε, σκιώδεις συγκητές. Ε, μπορείτε να είστε βέβαιος ότι εγώ τουλάχιστον θα το διαβιβάσω στον κύριο Πίπερ. Θα ήθελα να πληροφορήσω τον κύριο Τούρμες ότι η κυρία Φιώνα Χολ ε, και οι κύριοι Πίπερ και Τόμσεν δεν θα έρθουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό το ξέρουμε. Συνειδητοποίησαν. Um, Πάντως εγώ είχα καθήκον ως ηγητής να διευκρινιστεί αυτή η πληροφορία. Τώρα, αν ο καθένας για τους λόγους του κολλείεται να παραστεί στη συνεδρίαση. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου, πέντε λεπτά, πείτε μου. Και σταματήστε με αν, αν ξεπεράσω το χρόνο μου ή να βλέπω το χρονόμετρο, εν πάση περιπτώσει. Σημείο πρώτο. Από ό,τι ξέρω, η όλη συζήτηση ξεκίνησε πέρυσι τον Ιούνιο με την υποβολή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα χρόνο αργότερα ή ένα χρόνο και λίγες εβδομάδες αργότερα είμαστε πια σε θέση να πούμε ότι καταλήξαμε σε ευρία συμφωνία που την εστερνίζεται και το Συμβούλιο και αύριο επίσημα θα την ε, υπερψηφίσει και η Επιτροπή μας και η Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Οπότε η χαρμό συνείδηση είναι ότι παρά την δινή οικονομική κρίση η Ευρώπη λειτουργεί. Γιατί η θέσπιση τόσο περίπλοκη νομοθεσία μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σε ένα χρόνο περίπου, είναι ένα καλό παράδειγμα και μήνυμα ότι το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται για να δώσουν μια όθηση στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την αρχή θεώρησα ότι αυτή η νομοθεσία είναι μια πολύ σημαντική συμβολή, συνεισφορά για να διέλθουμε από την κρίση. Το 2000 ε, οι 27 χώρες μέλη που είναι σήμερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπάνησαν για τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου περίπου 50 και δισεκατομμύρια. Το 2011 οι ίδιες αυτές 27 χώρες δαπάνησαν περίπου 500 δισεκατομμύρια για την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Βέβαια, μειώθηκε αν το κοιτάσματά μας στη Βόρεια Θάλασσα και οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν στα ύψη. Ούτως ή άλλως υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα. Οπότε 500 δισεκατομμύρια ε, έφυγαν από την ευρωπαϊκή οικονομία με τέτοιου είδους νομοθεσίες προσπαθούμε να ανακτήσουμε, να φέρουμε πίσω ένα τμήμα τουλάχιστον αυτών των ε, τεράστιων νεκρών. Είναι ένα τεράστιο ε, έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου που έχουμε σε επίπεδο 27 χωρών μελών. Και με τέτοιου είδους νομοθετήματα θα μειώσουμε τις αγορές μας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και θα τι αντικαταστήσουμε από επενδύσει εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει περισσότερε θέσει εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο και θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε και κάποιες τεχνολογίες αποτελεσματικές αλλά και μοντέλα για να βοηθήσουμε τις βιομηχανίες μας να γίνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά. Όλοι μας χρειάζομαστε καινοτόμες τεχνολογίες για να μειώσουμε την ενεργειακή μας κατανάλωση στο μέλλον. Τώρα για την ίδια την οδηγία έχει δύο σημεία κυρίως. Τι είδους ε, ε, φιλοδοξίες υλοποιούμε με την οδηγία αυτή και ποια είναι η αρχιτεκτονική της. Να ξεκινήσουμε από την αρχιτεκτονική της οδηγίας. Ουσιαστικά μετατρέψαμε την πολιτική διακήρυξη του Μαρτίου του 2007 των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων που είπαν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ε, μειώσει κατά 20% τις εκπομπές και να αυξήσει κατά 20% την ενεργειακή απόδοση. Αυτή είναι μια πολιτική διακήρυξη σε συνεργασία με τα άρθρα 3 και 19. Εμείς μετατρέψαμε αυτή την πολιτική διακήρυξη σε ένα νομικό πλαίσιο όπου οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να αποφασίσουν για τους εθνικούς τους στόχους για την ενεργειακή απόδοση. Θα κοινοποιήσουν τους στόχους αυτούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 2014 θα προσθέσει όλα αυτά τα στοιχεία και αν το 2014 27 εθνικοί στόχοι δεν καταφέρουν να υλοποιήσουν αυτό το 20% τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση με νέα μέτρα για να ενισχύσει τους εθνικούς στόχους προκειμένου να υλοποιήσουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το 20% της ενεργειακής απόδοσης. Δεν θα μείνει λοιπόν ε, καινογράμμα η πολιτική διακήρυξη, αλλά θα λάβει σάρκα και οστά με αυτό το νομικό πλαίσιο. Έχουμε ένα σχετικά ασθενές άρθρο για τα δημόσια κτίρια, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά το αντάλλαγμα που λάβαμε, το αντικρίσμα ήταν ένα ισχυρό ε, άρθρο για ένα μακροπρόθεσμο οδικό χάρτη, ώστε να μπορέσουμε να εθετήσουμε όλες οι χώρες μακρόπνοες, μακροπρόθεσμες προοπτικέ για να μπορέσουν όλες οι χώρες να ανακαινήσουν ε, τα κτίρια τους. Άλλα σημαντικά άρθρα είναι το άρθρο 8 για τους καταναλωτές. Ε, το άρθρο 8 είναι ένα από τα άρθρα που δεν με ικανοποιούν πλήρω γιατί δεν δίνουν στους καταναλωτές όλα τα δικαιώματα που χρειάζονται και αξίζουν. Έχουμε άρθρα 13, ε, 14 και 15 πολύ καλά γιατί επιταχύνουν τις αγορές που ε, εξοικονομούν ενέργεια και προσπαθούμε να άρουμε εμπόδια και να διευκολύνουμε τις συναψυμβάσεων ε, όταν ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και αναγκάζουμε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τους εθνικούς τους κανόνες για, τις, για για τις ε, κατοικίες με πολλαπλή κυριότητα και πώς θα βελτιωθούν και στις περιπτώσεις αυτές τα θέματα της ενεργειακής απόδοσης. Τώρα, το σημείο 6 και ε, η υποχρέωση για 1,5 ενεργειακής οικονομίας. Αυτό ήταν επίμαχο κεφάλαιο. Τώρα ε, υιοθετήθηκε μία καταποκοπή εξαίρεση 25%. Λυπούμε, αλλά αυτό ήταν το τίμημα που χρειάστηκε να καταβάλουμε για να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι το αρνητικό. Το θετικό είναι ότι έχουμε έναν αντίκτυπο, γιατί θα έχουμε όλο και περισσότερες χώρες που θα αντιγράφουν την δανεική, γαλλική, αγγλική προσέγγιση για τις υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την ενεργειακή οικονομία. Ουσιαστικά οι εταιρείε που πουλούν σήμερα ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο στο μέλλον θα ενεργοποιούνται και στην αγορά υπηρεσιών ενέργειας. Και αυτό θα προσελκύει επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό των βιομηχανικών διαδικασιών που σήμερα ε, έχουν αποτελματωθεί γιατί δεν υπάρχουν αρκετές αποσβέσεις και αρκετά γρήγορη χρόνια επιστροφής. Είναι 12, 13 και παραπάνω μήνες. Αν λοιπόν οι ενεργειακές εταιρείες και οι βιομηχανίες ε, πυρώσει της προσπαθίες τους θα έχουμε πολύ πιο γρήγορη απόσβεση των επενδύσεων και ε, αποδοτικότητά τους. Επίσης, ε, το 2016 είπαμε ότι όλες οι εξαιρέσεις μπορούν να καταργηθούν γιατί θα έχουμε μια γενική αναθεώρηση της πρότασης. Και τέλος, τι επιτυχάνει η οδηγία ως προς τις φιλοδοξίες της. Ο στόχος όπως προβλέπει το άρθρο 3, είναι 20%. Η οδηγία σήμερα από μόνη της θα υλοποιήσει γύρω στο 15% Υπό τον όρο βέβαια, και αυτό με ανησυχεί κάπως, υπό τον όρο ότι θα έχουμε νέα οδηγία για το οικολογικό σχεδιασμό και την επισήμανση των boilers και θα συμπεριληφθεί σε αυτή τη γραμμή για το 15%. Και προβληματίζομαι γιατί μερικά κρατημέλη, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι και πολύ σαφή για το πότε θα ληφθεί υπόψη αυτό, η απόφαση για τον boiler. Ελπίζω να υιοθετηθεί αυτό το μέτρο και φυσικά το δεύτερο μέτρο που μπορεί να μας πάει πάνω το 15% είναι η νομοθεσία για το διοξείδιο του άνθρακα για τα οχήματα και τα λεωφορεία. Ίσως έτσι φτάσουμε στο 16,5% ίσως και 17%. Κάτι που σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο για το 20%. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα το 2014 θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τη ρήτρα αναθεώρηση του άρθρου 3 και το 2016 τη ρήτρα αναθεώρηση του άρθρου 6, ώστε να υλοποιήσουμε σίγουρα αυτό το στόχο του 20%. Και θα ολοκληρώσω με θερμότατες ευχαριστίες προς όσους ε, έλαβαν μέρος στην διαμόρφωση της έκθεσης, ιδιαίτερα στους και ηγητές, αλλά να συγχαρώ και την πρόεδρο, πρόεδρό μας, την κυρία Σαρτόρη, που πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και θερμότερες φυσικά ευχαριστίες προς το προσωπικό, τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες μας, τους βοηθούς μου, τον Φρανκ και τη Μισελ, αλλά συγχαρητήρια και στη γραμματεία, γιατί πραγματικά και ο Χάνες δούλεψε άοκνα όλη τη χρονιά και υπάλληλοι όλων των προσωπικών ομάδων και οι βοηθοί όλων των βουλευτών συνέβαλαν με την προσήλωσή τους και χάρη στη βοήθεια όλων αυτών καταφέραμε και διεκπαιρεώσαμε αυτή την οδηγία. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος όλων. Ο Βιντάλ Κουάδρας έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βεβαίως και είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή τη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον εισηγητή και όλους τους συμμετέχοντες, διότι Εργαζόμενοι ε, με την οδηγία αυτή για την ενεργειακή απόδοση φτάνουμε σε ένα παράδοξο. Η ενεργειακή απόδοση είναι ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος και πιο γρήγορος για να φτάσουμε στους στόχους μας σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια, μείωση εκπομπών και ούτω καθεξής. Συμφωνούμε απόλυτα όλοι ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μια πιο αποδοτική οικονομία ως προς τη χρήση της ενέργειας. Υπάρχει λοιπόν ομοφωνία ως προς το στόχο, ως προς το θέμα αρχής αυτή την Επιτροπή. Αυτή η οδηγία φτάνει σε μια δύσκολη στιγμή. γιατί απαιτεί από τις επιχειρήσεις του τομέα να καταβάλουν προσπάθειες μέσα στα πλαίσια μίας μακράς ύφεσης και οικονομικής κρίσης, μεγάλης οικονομικής κρίσης. Γιατί οι επιχειρήσεις όταν έχουν έναν επιπρόσθετο φόρτο τον απαρνούνται. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν και οι κυβερνήσεις πρέπει να μειώσουν το έλλειμμα, έχουν υψηλό χρέος, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Και τη στιγμή που προαπαιτείται μία νομοθετική πράξη και μία επενδυτική καθαρά προσπάθεια τις βρίσκει σε μια κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό το παράδοξο, από αυτή την αντίφαση. Νομίζω ότι ο Κλόντ μας είπε τι πρέπει να γίνει, να είμαστε ευέλικτοι. Η οδηγία ορίζει τους στόχους, ορίζει ορισμένες διαδικασίες και μεθόδους και παράλληλα αφήνει ένα περιθώριο ευελιξίας έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα και ανάλογα με τις συνθήκες, να μπορέσει να ανταποκριθεί αυτό που, αυτά που ορίζονται από την οδηγία. Γι' αυτό μιλάμε για ένα σοβαρό εγχείρημα ευθύνης και πιστεύω ότι στην πρώτη ανάγνωση φτάσαμε σε πολύ απτά και καλά αποτελέσματα. Θα πρέπει να συγχαρούμε και την πρόεδρο της Επιτροπής μας και την ομάδα του Κλοντ καθώς και την ε, γραμματεία της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας και Ενέργειας. Επίσης, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλή φόρμα και έτσι χάνουμε και περί τα κιλά. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Φιώνα Χολ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το προσωπικό που συμμετείχε σε αυτή την εργασία. Θα ήθελα να αναφερθώ στη Δανέζικη Προεδρία που διαδραμάτισε επικοδομητικό ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και τον Κλόντο Τούρμες, τον εισηγητή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να θυμηθούμε πώς φαινόταν αδύνατη αυτή η οδηγία για μεγάλο χρονικό διάστημα και θεωρήσαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να εντάξουμε 2.000 τροπολογίες σε ένα κείμενο, ε, κάτι το οποίο κατάφερε ο ίδιος. Φτάσαμε σε ένα κείμενο το οποίο διαπραγματευτήκαμε με το Συμβούλιο με την υποστήριξη των πολιτικών ομάδων. Μετά θεωρήσαμε ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο, γιατί η θέση μας βρισκόταν ε, πολύ μακριά, πήγε πολύ από εκείνη του Συμβουλίου. Γι' αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τον Κλοντ για τις δεξιότητές του και την ε, εμπιστοσύνη με την οποία ε, προώθησε την πίστη του στην οποία βασίστηκε για να προωθήσει αυτό το έργο. Φτάσαμε σε ένα πολύ καλό κείμενο κατά από δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι αν όλες οι διαπραγματεύσεις ήταν τόσο επιτυχείς, τότε θα ήμασταν ιδιαίτερα ευτυχείς όλοι. Ευχαριστούμε την κυρία Χόλ ο κύριος Τσίτσεστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λυπούμε γιατί έχασα ένα τμήμα της συζήτησης. Θα ήθελα όμως και εγώ να πω λίγα λόγια εκ μέρους της συναδέλφου Φόρτ που ζητά συγγνώμη για την απουσία της αλλά συμμετέχει κάπου σε ένα τριμερή διάλογο. Μου ζήτησε πάντως να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το πολύ αξιόλογο έργο του και να, να ευχαριστήσω και τους και εισηγητές γιατί ήταν πραγματικά μια συλλογική προσπάθεια, κοπιαστική, που είχε όμως πολύ αισιοπέρας. Νομίζω ότι όλοι αξίζουν συγχαρητηρίων για ένα πολύ δύσκολο και προβληματικό θέμα, επίμαχο, δεδομένου των τεράστιων διαφορών που υπήρχαν στην αρχή μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Η κυρία Φόρτ λοιπόν μου ζήτησε να πω ότι χαίρεται που η οδηγία θα προσφέρει στα κρατημέλη την δέουσα ελαστικότητα για να εφαρμόσουν μέτρα της ε, πολυπόθητης ενεργειακής απόδοσης. Ε, μερικοί συνάδελφοι λυπούνται για την ε, έλλειψη δεσμευτικών εθνικών στόχων. Δεν είμαι από αυτούς βέβαια που θλίβονται γι' αυτό. Η κυρία Φόρ θεωρεί ότι ε, ένας δεσμευτικό στόχο θα ήταν ε, λιγότερο αποτελεσματικό εθνικός από ότι τα δεσμευτικά μέτρα που υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει φυσικά ε, να αναλάβουν τις ευθύνε του και τα κράτη-μέλη. Φαίνεται ότι πρώτη φορά συμφώνησαν οι χώρε σε δεσμευτικέ υποχρεώσει για την ενεργειακή απόδοση. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάπως παρακινδυνευμένες αυτές οι δεσμευτικές υποχρεώσεις, αλλά εν πάση η κυρία Φόρντ, η σκιώδη συγκίτρια, θεωρεί ότι είναι ισορροπημένο το αποτέλεσμα, καλό συμβιβασμό και συγχαίρει όσοι συμμετείχαν στην διαμόρφωσή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίτσεστερ, κυρία Πιλάρντε Καστίγιο. Ευχαριστώ όταν ξεκίνησε η συζήτηση ήμασταν μόνο ο Κλώτ και εγώ. Δεν είχαν έρθει στο μεταξύ εκπρόσωποι των υπόλοιπων ομάδων. Στο μεταξύ γίναμε πιο πολλοί. Έλαβαν λόγο οι εκπρόσωποι όλων των άλλων ομάδων. Θα ήθελα να πω και εγώ εκ μέρους ομάδας μου και εκ μέρου του Μάρκου Πίπερ που ήταν ο σκιώδης συζητητή εκ μέρου του ΕΛΚ ότι και εκείνο αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που επιτελέστηκε σε συνεργασία με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους και εισηγητές και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για αυτό το πνεύμα συνεργασίας. Ως προς την ουσία, από ό,τι βλέπω εδώ στις σημειώσεις του σκιώδου συγητού, ο κύριος Πιπέρα θεωρεί ότι θα πρέπει, ε, μάλλον θα ελπίζαμε να δείξει μεγαλύτερη δέσμευση και μεγαλύτερη φιλοδοξία το Συμβούλιο. Τελικά το επίπεδο φιλοδοξίας του Συμβουλίου ήταν ε, χαμηλότερο από αυτό που περίμενε το ΕΛΚ. Πάντως, ο σκιώδης ηγητής μας παρόλα αυτά ε, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ε, οι υποχρεώσεις και οι φιλοδοξίες οδηγίες μπορούν να υλοποιηθούν με ελαστικό τρόπο, με ελαστικά μέσα. Η ελαστικότητα είναι σημαντικό στοιχείο για μας ε, και το λαμβάνουμε υπόψη προκειμένου να αποτιμήσουμε πολύ θετικά την οδηγία. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω. Είχαμε ήδη πολλές φορές, όπως σας είπα, την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πάντως, ε, η ομάδα μου ήθελε να ευχαριστήσει θερμά και να εκφράσει την έντονη υποστήριξη και της ομάδας αλλά και του Σκέδου του κ. Πίπερ για την έκθεση του κ. Τούρμες. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλοι εγγεγραμμένοι. Το λόγο λοιπόν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Επιτροπής θα ήθελα να σας πω και αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, αληθεύει ότι υπάρχουν κάποιες πτυχές που απογοητεύουν στο τελικό αποτέλεσμα. Θα συμμεριζόμαστε την ανάλυση όμως όλων εκείνων που ε, τοποθετήθηκαν στη συζήτηση ότι είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και δίνει τη βάση για να είμαστε αποτελεσματικοί με βάση μια αποτελεσματική πολιτική. Υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις που συγκεκριμένα και με σαφήνεια μπορούν να εντοπιστούν σε σχέση με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανέφερε τις ε, προοπτικές ε, για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ο κύριος Τούρμες και το αποτέλεσμα είναι καλύτερο σε σχέση με την αρχική μας πρόταση και αυτό χάρη στη δουλειά που έκανε το Ευρωκοινοβούλιο να διαπραγματευτεί και να υπάρξει αποτελεσματικότητα στις νέες ιδέες που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Χαιρόμαστε για την ευκαιρία. Κύριε Τούρμες, Πρόεδρε, και το σύνολο της ομάδας, της διαπραγματευτικής ομάδας ε, ήταν ένας αποτελεσματικός ε, και στεναρός εταίρος ε, για το Συμβούλιο και την Επιτροπή και γι' αυτό τον λόγο πετύχαμε αυτό το καλό αποτέλεσμα πιστεύω από τις Ευρωπαϊκές επιτροπή την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τρία πράγματα μπορώ να υποσχεθώ. Πρώτον, να ξεκινήσουμε με την υλοποίηση αυτής της οδηγίας με τα κράτη-μέλη άμεσα και δεύτερο, με υποθέτοντας ότι θα έχει ψηφιστεί προς έγκριση στην Ολομέλεια, θα πρέπει σε σχέση με τις ε, παλαιότερες ε, οδηγίες να ξεκινήσουμε σε σχέση με το Σεπτέμβριο να δούμε τι θα βρίσκεται επί τραπέζης. Δεύτερον, για το οικοσχεδιασμό θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα βαρύδια, τα, οποία, τα βάρη τα οποία ανέφερε ο κύριος ε, Τούρμες και να επιταχύνουμε την αναθεώρηση για να καλύψουμε τα κενά. Και τρίτον, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ήδη αναμένεται το 2014 να υποβληθεί η ανάλυση μας των εθνικών στόχων και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Ήταν μια αποτελεσματική εταιρική σχέση αυτή. Ευχαριστούμε για το ότι είχαμε μια τόσο καλή βάση για την εργασία μας. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Τούρμες για να συνοψίσει και να φτάσει να μας πει ορισμένα συμπεράσματα μετά από αυτή τη συνενετική διαδικασία. Νομίζω είναι εύκολο να ολοκληρώσουμε σε σχέση με αυτό το θελκτικό έτος και για μένα και τους κοιόδης και τους υπαλλήλους. Ήταν πραγματικά ελκυστικό το εγχείρημα. Είμαστε τώρα έτοιμοι να κάνουμε αυτές τις, ε, να έχουμε αυτό το διάλειμμα των θερινών διακοπών, να ανακτήσουμε την ενεργητικότητά μας μετά από αυτό το ευρύτερο πλαίσιο εργασιών που είχαμε φέτος και προσπαθειών μας. Αυτό που θα πρέπει να διασφαλίσουμε πιστεύω σε σχέση και με την ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι παρούσα και έκανε πολλή δουλειά και εκείνη. Όμως η περαιτέρω αναβολή των θεμάτων για τους ε, βραστήρες, θερμοσύφωνες ή βραστήρες ε, είναι κάτι που πρέπει να υπάρξει πίεση από την Επιτροπή στα κράτη-μέλη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για, γιατί διαφορετικά δεν ε, θα μπορούν τα πράγματα να βαίνουν σωστά. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι βραστήρες λοιπόν και θα πρέπει αυτό το πράγμα να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο. Και υπάρχει και μια δεύτερη πτυχή, όπου πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε σαφέστερα μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα δοθούν. Τη γραπτή δήλωση που διαπραγματευτήκαμε, e UTS, είχαμε μεγάλη μάχη που είχαμε δώσει για τον όρο κατεπήγων, urgent urgent κατεπήγον και μίλησα και με τον Πέτερ Λίζε από πλευράς εισηγητού της Επιτροπής Περιβάλλοντος που είναι και δόκτωρ. Όταν έρχεται κάποιος και αναφέρει ότι είναι κατεπήγον ένα θέμα, τότε ο γιατρός, ο δόκτωρας δεν παίρνει κάποιες διακοπές πρώτα εβδομάδων ή μηνών, προχωρεί αμέσω με τα αναγκαία μέτρα ή την εγχείρηση ο γιατρός. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι σαφέστατο ότι η γραπτή δήλωση που καταφέραμε να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η υπόσχεση που εντάσσεται στη γραπτή αυτή δήλωση, στην έγγραφη αυτή δήλωση για την αλλαγή εναλλακτικών λύσεων πρέπει να υποβληθεί και να λειτουργήσει πριν από το, τις θερινές διακοπές και όχι μετά. Διότι διαφορετικά θα υπάρξει εντύπωση που θα αποκομίσουν όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ουσιαστικά αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος, μέλος των διαπραγματεύσεων και με τη μείζωνα διαφορά που είχαμε με το Συμβούλιο ως προς αυτό, για τον τρόπο να πετύχουμε μια συμφωνία για την ETS, e ήταν η δυνατότητα αυτής της δήλωσης, δήλωσης και για θεσμικούς λόγους δεν είναι αποδεκτό μετά την υπογραφή αυτής της έγγραφης γραπτής δήλωσης το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ανταποκριθεί και να μην υλοποιήσει αυτά τα οποία υπέγραψε η ίδια. Δεν θέλω να είμαι πιο εξειδικευμένο και πιο λεπτομερή στι παρατηρήσει μου σήμερα, αλλά θα πρέπει να περάσετε στου ανωτέρου σα, στου προϊσταμένου σα, αυτό το μήνυμα από το Ευρωκοινοβούλιο. Τούτου λεχθέντος νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι πλέον να ψηφίσουμε προ έγκριση αύριο και με αυτόν τον τρόπο αυτή την πολιτική επιδόσεων και αποδοτικότητας που θα πρέπει και σε εθνικό επίπεδο να διοργανωθεί, όσο νωρίτερα καταλήξουμε και ξεκινήσει αυτή η δουλειά, τόσο το καλύτερο. Και γι' αυτό πραγματικά πιστεύω ότι πετύχαμε κάτι θετικό και για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών και επιχειρήσεών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τα πολύ καλά λόγια που ακούστηκαν από τον Τζάι στον Αλέχο Βιντάρ Πραγματικά τα εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά τα καλά λόγια. Σας ευχαριστούμε κύριε Τούρμες για άλλη μια φορά. Αύριο θα ψηφίσουμε. Αύριο προβλέπεται η ψηφοφορία. Λίγουν οι εργασίες της Επίτροπης. Θα συνεδριάσουμε αύριο στις 9 το πρωί. Τώρα αρχίζει η συνεδρίαση των συντονιστών. Έχουν ενημερωθεί για το ότι θα γίνει η συνεδρίαση αρκετά νωρίτερα.